την Προεδρία. Παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και σχετικά με τη διεθνή διάσκεψη για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στη Βενεζουέλα. Όπω γνωρίζετε, η ΕΕΔ μαζί με τον ΥΠΑ των Ηνωμένων Εθνών για του πρόσφυγε και τον Διεθνή Οργανισμό μετανάστευση. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στις Βρυξέλλες οργάνωσε διεθνή διάσκεψη για να κινητοποιήσει και να ενώσει τι ε, διεθνεί δυνάμει ε, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα. 4,5 εκατομμύρια Βενεζουέλ, Βενεζουελανών έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες σε μια από τις πιο δραματικές κρίσεις της εποχής μας ο αριθμός των ανθρώπων που διαφεύγουν από τη χώρα ε, θα μπορούσε να ε, ανέρθει σε 6,5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2020, κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ τα 5,6 εκατομμυρίων ανθρώπων που υπολογίζεται ότι έχουν εγκαταλείψει την Συρία μετά το 2011. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ότι η ανθρωπιστική αυτή κρίση είναι κρίση ανθρωπογενής που απαιτεί πολιτική λύση, μια δημοκρατική και ειρηνική λύση η οποία θα πρέπει να προέλθει από εντός της Βενεζουέλας και να την υποστηρίξουν η υπόλοιπη περιφέρεια και η διεθνή κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει εκφράσει την υποστήριξη του προς ε, την προσήλωση της κυρίας Μογκερίνη και πιστεύει ότι μόνο ε, ελεύθερες ε, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές μπορούν να αποτελέσουν μακροπρόθεσμη λύση για τη Βενεζουέλα. Θα ακούσουμε τώρα τον συνάδελφο Χαβιέρε Λόπε ε, που ήταν παρόν στη διάσκεψη αυτή και θα ακούσουμε και την κυρία Βερονίκ Λορένσο που είναι επικεφαλή του τμήματο για την Νότια Αμερική στην ΕΙΕΤ που θα μα ενημερώσει σχετικά με την ε, πολύ ευαίσθητη πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Θα μας παρουσιάσουν τα, αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της ε, Διεθνούς ε, Διάσκεψης Αλληλεγγύης της προηγούμενης εβδομάδας. Θα ακούσουμε επίσης ε, και τον κύριο Χόρχε Καπαλιέρα, που είναι επικεφαλής του, της Μονάδας για τη Λατινική Αμερική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Χαβιέρ Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως εξηγήσατε την περασμένη εβδομάδα 28 και 29 Οκτωβρίου είχαμε εδώ την Διεθνή ημέρα σχετικά με τους πρόσφυγες ε, της ε, Βενεζουέλα. Δεν θέλω να συμπληρώσω τα όσα είπατε, αλλά μόνο κάποιες σκέψεις σχετικά με τη συνάντηση αυτή, το συνέδριο αυτό και γιατί θα έπρεπε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή της ε, εκπροσώπου ώστε να φέρουμε στο προσκήνιο μια τεράστια κρίση, την μεγαλύτερη σε μέγεθος <coughs> στην ιστορία της Νότιας Αμερικής. 4,5 ε, εκατομμύρια που έχουν εγκαταλείψει τα, τα σπίτια τους ε, ε, αντίστοιχη ποσόστοση με μια πολεμική σύγκρουση. Και δυστυχώς εκτοπισμός, βίαιος εκτοπισμός, ο οποίος ίσως να μην είναι στην προσοχή της διεθνούς κοινότητας ε, όπως τα άξιζε. Η διεθνής κοινότητα που έχει και τις ευθύνε της. Η ανθρωπιστική κατάσταση δυστυχώς δεν έχει καμία τάση βελτίωσης, βράχη και μέσο πρόθεσμα. Ε, ε, τέτοιου είδους εκτοπισμοί απολύγουν σε νέες υποχρεώσεις και δημοσιονομικές για αυτούς που τους υποδέχονται. Το 80% εξ αυτών είναι στην περιοχή, στην Νότια Αμερική, στην Λατινική Αμερική, που αντιμετωπίζει δύσκολε κοινωνικέ καταστάσεις, δύσκολε πολιτικές καταστάσεις. Όλα αυτά απαιτούν πόρους σε πολύ βεβαρημένου ήδη προπολογισμού κρατικού, ε, Η διαδικασία του Κίτο προκειμένου να διοργανωθεί και να συντονιστεί η πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, στην ε, έλλειψη αναγνώρισης ε, πτυχίων, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι περίπλοκες και που οδηγούν σε εκτοπισμούς ε, τεράστιες κλίμακας όπως έλεγα. Εμείς παρενεύουμε στο συνέδριο, εγώ το έκανα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ήθελα να σημειώσω ότι αναφέρθηκαμε στα θύματα, αναφέρθηκαμε στις χώρες υποδοχής, στην Κολομβία, το Εκουαδόρ, το Περού και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Αναφερθήκαμε στην ανάγκη συνέχεια συνεργασίας και, οικονομικά δηλαδή σε επίπεδο διεθνού κοινότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Και πολύ σύντομα, καταρχάς εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πολύ προσεκτικοί. 11 ψηφίσματα από το 2014 έχουμε κάνει. Αυτό είναι θετικό και είναι καλό. Μάλλον δεν εστιαστήκαμε επαρκώς στις συνέπειες. Συνέπειες ανθρωπιστικά τη κρίση αυτή και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σε επόμενους μήνες και στην Ολομέλεια να εστιαστούμε πιο προσεκτικά ακόμα στις συνέπειες αυτές, ιδιαίτερα για κάποιες χώρες περιοχής. Και ήθελα επίση να θυμίσω ότι η λύση για τη χώρα που είναι η μόνη εγγύηση σταθερή λύση στο φαινόμενο αυτό θα έπρεπε να είναι ειρηνική, δημοκρατική που να ασκήσει πίεση στο καθεστώς που αυτή τη στιγμή ασκεί τον κρατικό έλεγχο, λέει ο μιλητής στη Βενεζουέλα, γιατί βρισκόμαστε σε μια ατραπώ χωρί διέξοδο αυτή τη στιγμή με θύματα του ανθρώπου. Σα ευχαριστούμε κύριε Λόπε, για την ενημέρωση και τα συμπεράσματα σας από τη διάσκεψη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βερονίκ Λορέντσο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που καλέσατε την ΑΕΤ στην ανταλλαγή αυτή απόψε. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Λόπες. Όντως, Βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο στη Βενεζουέλα και οι συνέπειες του είναι τραγικές, οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές και φυσικά τεράστιες επιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζουν την σταθερότητα της περιοχής. Να σας δώσω μερικά στοιχεία. Γνωρίζετε ότι έχουμε 7 εκατομμύρια Βενεζολονούς που χρειάζονται βοήθεια. Πάνω από 90% του πληθυσμού ε, διαβεί κάτω του κατοφλίου ποιότητα. 3,7 ε, εκατομμύρια ποσιτίζονται κάτω από φτώχεια και πάνω από το 70% των παιδιών δεν πηγαίνει σχολείο. Επίση, 5.000 ε, άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα μέρα με τη μέρα, καθημερινά. Και έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Και μάλιστα έχουμε βαθύτατα θεσμικά προβλήματα, συνεχής διάβρωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα αυτή. Επίσης, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναφέρει η Μισελ Μπασιλιέ, η πατή εκπρόσωπος των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με πολύ σοβαρό, σοβαρούς ε, ισχυρισμούς που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Βέβαια, η Βενεζουέλα έχει εκλεγεί ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει την υποχρέωση ως τέτοιο μέλος να προωθήσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνεργαστεί με τις ιδιαίτερες διαδικασίες και μηχανισμούς του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένες και μιας διερευνητικής αποστολής που στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια συστημική κρίση και σίγουρα δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε την κρίση, να την αντιμετωπίσουμε χωρίς δημοκρατικές εκλογές, χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου και την ε, επαναφορά ενός ανεξάρτητου συστήματος ελέγχων και ισορροπιών. Μας προβληματίζει ε, και η ε, ανάκληση των δύο διαμεσολαβητών από την Ορβηγία και φαίνεται ότι η διαδικασία δεν έχει την απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα. Θα πρέπει η μετάβαση να γίνει συνενετικά με εκλογές προεδρικές και με την εξασφάλιση εχεγγύων θεσμικών που θα επιτρέψουν μια πολιτική συνύπαρξη. Και παρόλο που η λίστα πρέπει να δοθεί αποκλειστικά από τη Βενεζουέλα, τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε ότι το εύρος, η εμβέλεια της κρίσης και οι γεωπολιτικές ε, ε, επιπλοκές της ε, χρήζουν ενεργό υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και συνεργασία με συμπληρωματικότητα ώστε να στηρίξουμε μια ειρηνική επαναφορά στη δημοκρατία και στην συνταγματική τάξη στη συνταγματική ένωμη τάξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Διεθνούς Ομάδας Επαφής συνέχισε να δίνει έμφαση στη διπλωματία προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό περιθώριο και είμαστε κατά των δύο λύσεων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω πόλωση και σε επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Είχαμε μάλιστα μια συνάντηση των υψηλόβαθμων ε, στα πλαίσια της ομάδας ε, συνδέσμου ε, παράλληλα με την διάσκεψη της περασμένης εβδομάδας και η διακήρυξη των εμπειρογνωμόνων επικρίθηκε δρυμύτατα από το καθεστώς της Βενεζουέλας. Θα πρέπει τώρα να συνεργαστούμε με τους ε, με διεθνείς παράγοντες και να συνεχίσουμε τις ε, στενές επαφές με εθνικούς ε, φορείς στη Βενεζουέλα. Επίσης έχουμε τον κύριο Ιγλέσιας που είναι ο ειδικό απεσταλμένος για τη Βενεζουέλα και θα μεταβεί στο Καράκας στο έγκυς μέλλον. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να επισημαίνω για την πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ότι συνεχίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκούμε πιέσεις και μέτρα πίεσης προς τη Βενεζουέλα. Και αν οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφορήσουν και δεν γίνουν καλοπροαίρετα, τα μέτρα θα παραμείνουν ενισχύ. Είναι βέβαια στοχευμένα μέτρα, δεν θα επηρεάσουν τον πληθυσμό και επίσης είναι αναστρέψιμα εφόσον διαπιστώσουμε κάποια πρόοδο. Μάλιστα έχουμε ε, στις 26 Σεπτεμβρίου υιοθετήσει νέε κυρώσει για 7 συγκεκριμένου ιδιώτε, ιδιαίτερα μετά από το θάνατο κάποιου. Και έχουμε 25 τελικά ιδιώτες που είναι αντικείμενο των κυρώσεών μας. Και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση σε περίπτωση που διακοπούν οριστικά οι διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό σκέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, από το 2018 παράσχει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 170 εκατομμύρια ευρώ έχουμε προσφέρει και εντός της Βενεζουέλας και στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα έχουμε προοδευτικά ενισχύσει τις δεσμεύσεις μας προκειμένου να βοηθήσουμε τους κατοίκους της Βενεζουέλας και εντός της χώρας αλλά και να βοηθήσουμε τις γειτονικές χώρες που προσπαθούν να, ε, να στεγάσουν τους, ε, τα, τα εκατομμύρια των προσφύγων και μεταναστών. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του ΚΙΤΟ, ε, η διαδικασία αυτή ε, ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να εναρμονιστούν οι πολιτικές και οι διαδικασίες και να αντιμετωπιστεί ε, συνολικά η κρίση. Βέβαια, η κρίση αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες ε, από τις χώρες της περιοχής. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ε, δεν ε, βρέθηκε στο επίκεντρο των δικών μας προτεραιότητων. Γι' αυτό και ήταν υποχρηματοδοτούμενη βέβαια είναι από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής και μέχρι τα τέλη του έτους θα γίνει από τις σημαντικότερες κρίσεις παγκοσμίω η κρίση της Βενεζουέλας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε ε, ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά και να προβλέψουμε τα κατάλληλα κονδύλια για να ελαφρύνουμε τις γειτονικέ χώρες της Βενεζουέλας που έχουν υπομειστεί όλο το βάρος ε, της μαζικής ε, μετανάστευσης. Γι' αυτό και συγκαλέσαμε την περασμένη εβδομάδα την Διεθνή Διάσκεψη Αλληλεγγύης, τη ιδιοργανώσαμε με την Ήπατη Αρμοστία και την Διεθνή Οργάνωση για τη Μετανάστευση. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας ε, συνοψίσω τα συμπεράσματα της διάσκεψης. Ήταν πολύ επιτυχημένη από άποψη συμμετοχής, από άποψη προβολής, αλλά και από άποψη ουσίας και περιεχομένου. 120 αντιπροσωπείες συμμετείχαν ε, με 500 μέλη συνολικά στη διάσκεψη αυτή και είχαμε 15 ε, υπουργούς. Ήταν καλή και κάλυψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και στον τύπο και παρουσία έντονη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε μπορώ να πω ότι ο στόχος μας υλοποιήθηκε, δηλαδή έγινε ευαισθητοποίηση της κατάστασης. Είναι πραγματικά δεινή κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών της Βενεζουέλας. Πλέον ο κόσμος το συνειδητοποίησε. Και επίσης κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου. Αν δεν βρεθούν εφάνταστες λύσεις, η κατάσταση θα εκφύγει το ελέγχου και θα γίνει ακόμη πιο τραγική. Θα ήθελα να σταθώ και σε τρία σημεία ως προς το περιεχόμενο των συζητήσεων. Τρία ήταν αυτά που αναδείχθηκαν. Καταρχήν, η ανάγκη συλλογική δράσης Αναφέρθηκα ήδη στη διαδικασία του Κίτο. Είναι σημαντικό οι χώρες αυτές, οι γειτονικές χώρες, να εναρμονιστούν στην αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών, όχι μόνο για να μετριάσουν τα, την ανθρώπινη οδύνη, αλλά για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ελαφρύνουν το βάρος των διοικήσεών τους. Βέβαια η πίεση συνεχίζεται γιατί η έξοδος των Βενεζολών συνεχίζεται. Επίσης υπάρχουν εντάσεις και ταυτόχρονα αυξάνεται η ξενοφοβία όσο εντείνεται αυτή η μαζική έξοδος ε, των κατοίκων της Βενεζουέλας. Γι' αυτό και θα χρειαστεί να στηρίξει τις χώρες αυτής της διεθνής κοινότητα. Επίσης τα ανθρωπιστικά μέτρα θα πρέπει να τις συνδυάσουμε με τις την ικανοποίηση των μακροπρόθεσμων αναγκών ε, ένταξης, κοινωνικής ένταξης των μεταναστών η κρίση αυτή όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά θα επιδεινωθεί πριν ξεκινήσει μια βελτίωση. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία προοπτική των κατοίκων τη Βενεζουέλα για επαναπατρισμό, για επιστροφή στι αιστείε του. Πολλέ χώρε μίλησαν για την ανάγκη να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, ώστε να συμβάλλουν οι Βενεζουελινοί στην οικονομική του ανάπτυξη. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε δημιουργικές εφάνταστε λύσει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης, ίσως ε, να προσελκύσουμε και ιδιωτικά κονδύλια και επενδυτικές τράπεζες για να μοχλεύσουμε ε, τα κονδύλια των δωρητών. Πραγματικά σοκαρίστηκα στις θεματικές ενότητες της διάσκεψης από το πόσο ε, το μέγεθος της οδύνης κυρίως γυναικών και παιδιών. Ε, τι έκθεση είχε η βία εις βάρος των γυναικών και πώς έχουν πληγεί οι άμαχοι. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους και κονδύλια, γιατί όσο ε, συνεχίζεται η έξοδος, ε, όλο και πιο βάλλοντα τμήματα του πληθυσμού θα πέφτουν στα δίχτυα κυκλωμάτων διακίνησης και θα είναι θύματα ξενοφοβίας και καταχρήσεων. Η περιορισμένοι πόροι που έχουμε μέχρι στιγμή ε, έδειξαν την ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτέ τι πιο ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού. Επίση, η διάσκεψη αυτή δεν ήταν διάσκεψη δωρεών. Παρ' όλα αυτά έγιναν κάποιε υποσχέσει δωρεά που ανέρχονται συνολικά σε 120 εκατομμύρια ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, επιβεβαίωσε τις, ε, τη δέσμευσή της να διατηρήσει αμύωτο το επίπεδο υποστήριξης που έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Επίσης, ε, δεν αρκεί αυτή η διάσκεψη. Θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα συστηματικών προσπαθειών για την κινητοποίηση περισσότερων κονδυλίων. Θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Έχουμε τη συνάντηση του, στην Ποκοτά τον, στα μέσα Νοεμβρίου της διαδικασίας του Κίτο. Επίσης, στα μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε μια πρωτοβουλία. Στο Κίτο επίσης ε, μια εκδήλωση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Και ίσως θα μπορούσαμε να συγκαλέσουμε και μία διάσκεψη για υποβολή δωρεών ε, στο πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους. Ίσως ε, στο περιθώριο της συνάντησης της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο στη Βόσιγκτον. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε λίγα λεπτά ακόμα, χωρίς διερμηνία, όμως αποκλειστικά στα αγγλικά. Δίνω το λόγο, το λόγο στον κύριο Καβαλιέρα. Παρακαλώ να είστε σύντομος δύο λεπτά. Thank you, Mr. Chair. I was planning to speak in Spanish. Let's switch into English. Um, anyway, I think the Commission shares the point of view expressed by those who took the floor before us